να συνεχίσω τη συζητήση επί των θεμάτων τους επόμενους μήνες και χρόνια. Να συζητάω μαζί σας δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για να κλείσουμε τη συζήτηση. Έχουν το λόγο και πάλι δύο λεπτά ο κάθε εισηγητή. Καταρχήν κυρία Σαϊφή έχει το λόγο. Euh,